με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού αν δεν υπάρχει αντίρρηση ο κύριος ε, Κούλοκλο ε, θα έχει έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφού δηλώσει ότι ε, δεν έχει κάποια θέση που να είναι συμβίβαστη. Τώρα η ομάδα ECR μου ζητά να διοριστεί ο κύριος Άμσατ Μπασίρ ως μέλος της για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν. Υπάρχουν παρατηρήσεις, όχι από ό,τι φαίνεται, οπότε ο διορισμός αυτός εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε την προφορική ερώτηση στην Κομισιόν, μηδενική ενοχή για τον ακροτηριασμό των γυναικών.